Ξεκινάει και γίνεται επανάληψη της συνόδου. Σας παρακαλώ να καθίσετε. το πρωτόκολλο της συνεδρίασης της 1 και 2 Φεβρουαρίου και τα εγκεκριμένα κείμενα τα έχετε λάβει. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις θεωρούμε ότι τα πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται ούτως.